Ε, εάν απειλείται το πρόγραμμα Έρασμους Και θα δώσω και πάλι το λόγο στον ε, Υπουργό Ανδρέα Μαυρογιάννη εξ ονόματος του Συμβουλίου. Υπουργέ, το μικρόφωνο, αν έχετε την καλοσύνη. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κύριε Κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτισμού, κυρία Πακ, αξιότιμα μέλη, Επίτροπε. Το Συμβούλιο συμμερίζεται απολύτως την άποψη ότι οι ε, οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης εξαρτώνται πάρα πολύ από το ανθρώπινο δυναμικό που θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο, μορφωμένο και με προσόντα. Και το πρόγραμμα διαβίου μάθησης συμπεριλαμβανομένου και το του των είναι από τα πιο επιτυχημένα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της παιδείας. Γι' αυτό τον λόγο επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι χρηματοδότηση ε, του προγράμματος διαφύου μάθησης για την περίοδο 2012-2013 δεν θα διακυβευθεί. Σε ό,τι αφορά το 2012, το Συμβούλιο άρχισε να αναλύει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχουν ε, ε, προταθεί στο σχέδιο τροποποίησης του προπολογισμού υπαριθμών 6 και το συντομότερο θα εγκριθεί σε ό,τι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων για το 2013, αυτές θα αποφασιστούν από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης ε, διαπραγμάτευσης για τον προπολογισμό. Είμαι πεπισμένος ότι και τα δύο σχέλη της Δημοσιονομικής Αρχής θα καταλήξουν σε ισορροπή συμφωνία το Νοέμβριο για τον προπολογισμό του 2013, όπως προβλέπει η συνθήκη. Τέλος, σε ό,τι αφορά το μέλλον του προγράμματο διαβίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένου προγράμματο Έρασμο, γνωρίζετε όλοι ότι οι διαπραγματεύσει που αφορούν ε, το επόμενο πολιτείας δημοσιονομικό πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι ακόμα εν εξελίξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέχεται στι διαπραγματεύσεις αυτέ. Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, Αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν σωστό να σας πω περισσότερα, διότι θα πρέπει να περιμένουμε την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ και εγώ, ε, Υπουργέ, και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι, εξ ονόματος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, πρόσφατα Ακούστηκαν πολλές εικασίε και πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τη μοίρα του Εράσμού. Πολλές εικασίε και στα μέσα μαζικής ενημέρωση, πολλέ αβεβαιότητε. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν χαίρεται που μπορέσει τώρα να διευκρινίσει τα... του θέματος αυτού. Είναι καθήκον μου να αναφερθώ στο Εράσμους μέσα στο συνολικό πλαίσιο έλλειψης χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που δεν αφορά το έρασμος μόνο. Το έρασμος είναι ένα τμήμα του προβλήματος. Ένα μικρό τμήμα του προβλήματος, αλλά πολύ ορατό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το 2012. Αυτό οφείλεται στην ε, συστηματική ε, υπο, στο συστηματικό ε, προϋπολογισμό που κάνουμε προς τα κάτω. Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε σωστό προϋπολογισμό και απέναντι στους πολίτες και προς τα έξω. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε ένα διορθωτικό προϋπολογισμό για φέτος. Ένα μεγάλο ποσό για την συνοχή και την ανάπτυξη πέθρου, αλλά και για τις εξωτερικές μας υποχρεώσεις καθώς και για τον τίτλο 1α που αφορά την ανταγωνιστικότητα και που καλύπτει ε, πολλά ερευνητικά προγράμματα που συμπεριλαμβάνει και το πρόγραμμα διαβίου μάθηση, ε, του οποίου είναι τμήμα το Εράσμους. Το lifelong learning, δηλαδή το πρόγραμμα διαβίου μάθησης αφορά και την δυνατότητα που έχουν οι ενήλικες για μάθηση, ε, αφορά και την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, αλλά το πιο ε, λεπτό και ευαίσθητο τμήμα είναι η κινητικότητα των φοιτητών, το εράσμος δηλαδή. Για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίε που είχαμε φέτος, ε, πρέπει να βρούμε 6 ε, εκατομμύρια ευρώ. Για ε, το lifelong learning χρειαζόμαστε 180 εκατομμύρια για όλη τη χρονιά. 90 εκατομμύρια χρειαζόμαστε για το Erasmus περίπου. Η δέσμευσή σας για την πρόθεση της επαγγελματικής ε, κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Γιατί παράλληλα με τα ετήσια προβλήματα, αυτό που διακυβεύεται είναι και το μέλλον του προγράμματος αυτού. Το πρόβλημα αυτό όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στις, και στις διαπραγματεύσεις για το πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020. Ε, θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τη θέση της εκπαίδευσης. Θα πρέπει νέοι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν το σωστό μείγμα ε, γνώσεων για να ξεφύγουν από το φάσμα της ανεργίας. Ε, επομένως, το μέλλον του, αυτό που, αυτό που ονομάζουμε Erasmus for All, αυτό είναι ένα από τα διακυβεύματα. τώρα όμως πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το Erasmus 2012-2013. Ε, ένα συνάδελφό σα ε, έκουσε τον κόδωνα κινδύνου για το Εράσμου για φέτο. Και 99% ε, αυτό που, αυτό που έχουμε στην τσέπη μας, δηλαδή τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, έχουν ήδη δοθεί στου εθνικού εθνικούς οργανισμούς στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε επαφή μαζί μας όχι μόνο οι εθνικοί οργανισμοί πληρωμή, αλλά έχουμε 33 συμμετέχουσες χώρε ε, συνολικά η Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, Κροατία και Ελβετία συμμετέχουν επίσης. 99 αυτών που είχαμε στη διάθεσή μας για το 2012 έχουν ήδη καταβληθεί στους εθνικούς οργανισμούς, ε, που είναι 33 εν το σύνολο τους. Έχουμε ήδη αιτήσει για φέτο, για 160 εκατομμύρια. Περιμένουμε και, άλλες, και άλλα αιτήματα να καταφτάσουμε στο 2012 είναι εύκολο να λέμε ποιο δεν θέλει ε, επιπλέον λεφτά. Βουλγαρία, Ρουμανία, Πορτογαλία κτλ. Οι υπόλοιπε χώρες ε, που στέλνουν αιτήματα για επιπλέον χρήματα είναι όλες οι υπόλοιπε και η διόρθωση του φετινού προπολογισμού είναι απαραίτητη. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα φέτος περισσότερα χρήματα. 180 ε, εκατομμύρια επιπλέον. Τα μισά είναι για το Εράσμου, τα 90 εκατομμύρια. Ο ε, Υπουργό ο κ. Μαυρογιάννη έχει δίκιο. Ε, είναι το καθήκον μας να εφαρμόσουμε σωστά το Εράσμους ε, το 2012 και στι αρχέ του 2013. Έχουμε ήδη προκαταβάλει στους εθνικούς οργανισμούς πολλά λεφτά. Αλλά αν δεν μας μείνει τίποτα, αν δεν προκύψει, αν δεν έλθει τίποτα άλλο, θα έχουμε πολλαπλά συσσωρευμένα προβλήματα το 2013. Γιατί τα πανεπιστήμια δεν θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των φοιτητών και θα μειωθεί η κινητικότητα των φοιτητών μέσα στο 2013. Γι' αυτό ακριβώς σας ε, καλώ, κάνω έκκληση και κάνω έκκληση και προς την Προεδρία να κάνετε ό,τι μπορείτε ούτω ώστε να υπάρξει σημαντική αύξηση 2012, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτή την σώρευση των προβλημάτων σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, το 2013. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Θα δώσω πρώτα το λόγο στη συνάδελφο Ντόρι Πάκ εξ του ΕΛΚ. Κύριε Προεδρεύον, <clears throat> κύριε Επίτροπε, Κύριε Προεδρεύον, σας άκουσα προσεκτικά, αλλά δεν σας πιστεύω. Γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Αποτυχία. Ομολογία αποτυχίας για τις αρμόδιες κυβερνήσεις, όχι του Κοινοβουλίου ούτε της Επιτροπής. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν πρόκειται για αύξηση των κονδυλίων επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δούλεψε πλημελώς, το μόνο ε, που θέλουν ε, που πρέπει να γίνει είναι ότι οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί ε, δεν σέβονται τις ε, υποχρεώσεις τους απέναντι στους νέους. Τα λένε όλα αυτά πόσο σημαντικά είναι την Κυριακή σε διάφορες ομιλίες για την κοινωνία. Είναι σημαντικό να κυκλοφορούν Και με την Πολόνια ήδη τους έχουν δυσκολέψει τη ζωή και τώρα αυτή η ναυαρχίδα, αυτό το σύμβολο που λέγεται αερασμός πλήττεται. Είναι γεγονός ότι και με τον ερασμό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους νέους ε, η διαμονή στο εξωτερικό και δεν μπορούν καν να βασιστούν στις δεσμεύσεις των πολιτικών. Αυτό είναι ολέθριο μήνυμα, ιδιαίτερα για εκείνους που χρειάζονται επιγόντως τη χρηματική στήριξη στον έρασμο. Επανειλημμένα οι Υπουργοί Παιδείας έχουν ε, διατρανώσει και τώρα το ξαρακούμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε στο στόχο μας για το 2020 να μπορούν πολλοί νέοι να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να διαμένουν εκεί. Μα ούτε το 5% των φοιτητών δεν μπορούν να πάνε στον έρασμο γιατί το ταμείο είναι μείον. Ε, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου δεν θα πρέπει να ε, εξοικονομούν χρήματα στην πλάτη των φοιτητών. Εκεί θα πρέπει να δείχνουν μεγαλοψυχία γιατί πρόκειται για το μέλλον και των δικών τους παιδιών. Thank you very much. Ευχαριστώ. Όταν σπούδασα στη Βιέννη, εγώ δεν είχα την ευκαιρία τότε να επωφεληθώ από το Εράσμος και λυπάμαι ακόμα που δεν είχα αυτή την ευκαιρία. Τώρα πολλοί νέοι στην Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα, την έχουν ακόμα πρέπει να πω, γιατί και αυτό ακόμα ε, είναι σε κίνδυνο για κάποιους νέους. Στην Ευρώπη μιλούμε για την ανάγκη αριστείας υψηλών προσόντων, γλωσσομάθειας. Το πρόγραμμα Εράσμους απειλείται όμως. Στην Ευρώπη όλοι οι ηγέτες μιλούν για την ανάγκη κινητικότητας. Δεν μπορούμε να μένουμε προσιλωμένοι σε ένα τόπο, σε μια χώρα. Και ορισμένα κράτη-μέλη ε, απειλούν την κινητικότητα. Άλλος μιλάει για μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που θα πρέπει να, έρθει, να προσθεθεί στην εθνική μας ή στην τοπική μας ταυτότητα. Και πάλι ορισμένοι ηγέτες απειλούν ε, και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι ορισμένες από τις χώρες που θέλουν πολλοί ε, φοιτητές να πάνε στον έρασμο προσπαθούν να κόψουν τον προπολογισμό, να τον περιορίσουν. Και αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Συμφωνώ πολύ με τα λεγόμενα του Επιτρόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, και σας κύριε Μαυρογιάννη. Είστε πάρα πολύ ευγενείς και προσινείς ε, και καλός, αλλά καμιά φορά να δείχνετε λιγότερη καλοσύνη απέναντι στους συναδέλφους σας των άλλων κυβερνήσεων, γιατί είναι αδύνατα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Ε, και είναι ναυαρχίδα το χαρακτήρισε η κυρία Πακ αυτό το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ταυτότητας Συνάντησης. Ε, είμαστε οι πιο κατερτισμένοι και εκπαιδευμένοι στην Ευρώπη. Και τέτοιους καιρούς τώρα ερχόμαστε να τα απειλούμε όταν αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμό. Λέμε στου νέου θέλετε να είστε πραγματικοί Ευρωπαίοι, λυπόμαστε, αλλά λεφτά δεν έχει για αυτή την υπόθεση. Ε, καμιά φορά θα πρέπει να είστε πιο σκληρός απέναντι στους συναδέλφους σας κύριε Μαυρογιάννη και να τους λέτε τι λέει το Κοινοβούλιο και μάλιστα ομόψυχο. Χρειαζόμαστε τον έρασμο και με επαρκή χρηματοδότηση για τους νέους, γιατί πρόκειται για την Ευρώπη και όχι για τις εθνικές τους φιλοδοξίες. Ευχαριστώ. Thank you very much, President. And our colleague... Ευχαριστώ. Λόγο στον κύριο Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για όλα όσα είπατε. Έχω να σχολιάσω κάποια πράγματα κι εγώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου συνηθίζουμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας, έτσι, δεν το συζητάμε το θέμα αυτό. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτή τη συζήτηση για τις συνέπειες του μειωμένου προϋπολογισμού που ανέφερε ο κύριος Επίτροπος. Βρισκόμαστε σε μια συζήτηση παράλογη. Οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν καθόλου αυτή τη λογική. Όταν υπάρχουν λογαριασμοί θα πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι λογαριασμοί θα πρέπει να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας, γιατί αυτό μειώνει την αξιοπιστία μας. Αν δεν σεβαστούμε τις υποχρεώσεις μας, νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και αυτό είναι και ευθύνη των κρατών μελών. Και δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τους φοιτητέ αυτή η ιστορία. Τους ξεπερνάει το πρόβλημα των φοιτητών. Οι φοιτητέ είτε δεν θα βοηθηθούν, θα μειωθεί η βοήθεια που του δίνεται πάντω. Πάντω τα πράγματα δεν είναι καθόλου αφηρημένα, είναι πολύ απτά. Πολύ απτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και αυτά συζητάμε. Και εδώ σα κάνω, σα κρούω τον κόδωνα. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ε, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να γίνει όμοιρος σε, μια, σε ένα παιχνίδι τακτικής ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να αποφύγουμε οι νέοι να τους χρησιμοποιήσουμε τελικά ως πειραματόζωα και ως ε, ε, ομήρους. Θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ δημοφιλές. Όλοι το ξέρουν, όλοι το καταλαβαίνουν. Είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό διακυβεύεται. Δεν μιλάμε τώρα για ευρώ και για πεντάδεκάρες ε, τόσα πάνω τόσα κάτω. Κάνω σύσταση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, ούτω ώστε αυτό το πρόγραμμα να έχει επαρκή πόρους. των Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου, αξιότιμη κύριε Επίτροπε Λεβαντόφσκι. Ναι, δυστυχώς είναι σωστό αυτό. Σήμερα ανακαζόμαστε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι ικτρή η κατάσταση στο πρόγραμμα Εράσμος. Οι φοιτητέ δεν έχουν πια τα χρήματα για τις υποτροφίες που τους είχαν υποσχεθεί. Είναι τελείως αντιφατικό με τους στόχους και πρέπει να αποταθώ σε εσά, κύριε εκπρόσωπε τη Κυπριακή Προεδρία, στου στόχου που το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο αποφάσισε, δηλαδή περισσότερα για τον έρασμο, περισσότερα για την κινητικότητα των σπουδαστών και των φοιτητών, περισσότερο για την παιδεία και τη μόρφωση των νέων μα. Πώ μπορεί κανεί να είναι τόσο ανεύθυνο όσο και μείοψ και να μην ε, μπορεί να συνεχίσει από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα, το πρόγραμμα Έρασμος, να κλείνεται τον κρουνό τη χρηματοδότηση Πολύ σωστά είπε η κυρία Πακ. Ήδη έχουμε εφαρμογή 99% από τον Οκτώβριο. Τι θέλουμε περισσότερο. Αν θέλετε να κάνετε οικονομίες, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις για τον καπνό, που κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά και όχι για ένα τέτοιο πρόγραμμα που μόνο όφελο σημαίνει για τους συμμετέχοντες, όλους. Παραβιάσατε τη συνθήκη, διότι δεσμευτήκατε για ανάληψη υποχρεώσεων που δεν τιμάτε. Και αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δυστυχώς ε, κατά συνέπεια την αξιοπιστία της σύνολης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι βαρύ πολιτικό σφάλμα. Και δεν είναι μόνο αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα εράσμους, αυτή η αυαρχίδα που πιέζεται, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που είναι επίση μείον ξέρετε τι κινδυνεύεται και να μην υπάρχουν χρήματα για ε, προγράμματα καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και της μακροχρόνιας ανεργίας. Αυτό είναι τελείως αντιπαραγωγικό από αυτά που εξαγγέλλεται πάντα στις συνόδους κορυφής για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ότι θα πρέπει λένε, θα του τους νέους στην Ευρώπη να μετακινούνται, να ταξιδεύουν, να εμπλουτίζουν, να μεταμορφώνονται. Σταματήστε επιτέλους αυτή την ανεύθυνη πολιτική να εγκρίνουμε έναν ε, διορθωτικό προπολογισμό και με θάρρος να πάμε στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί πραγματικά αυτά τα χρήματα χρειάζονται για την παιδεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι η κυρία Πάκ, ο κύριος Βόμποντα, ο Δανός συνάδελφος, όλοι ανησυχούν. Και οι ανησυχίες αυτές είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Αυτά που είπατε μας τάραξαν, γιατί είναι ένα πρόγραμμα που αξίζει να του δοθούν κονδύλια και να γίνουν επενδύσεις. Η κυρία Τρούπελα εξέφρασε τις ανησυχίες της επίσης. Και είπε, συχνά κατασπαταλάμε χρήματα, αλλά τα χρήματα που δίνουμε για το έρασμος δεν είναι σπατάλη, είναι επένδυση. Και όλοι μας, και ειδικά η Επιτροπή, αλλά και το Συμβούλιο, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν ε, χρήματα στον κουμπαρά του Εράσμους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι φοιτητέ που σπουδάζουν στην Πολωνία παίρνουν πολύ περισσότερα του Πολωνού που σπουδάζουν στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Αυτό είναι λάθο. Δεν πρέπει να παίρνουν όλοι τα ίδια. Το βασικό είναι όμω να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν χρήματα. Δεν τελειώνουν τα χρήματα. Δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο, στου πολίτε μα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί αυτή την αυαρχίδα, αυτό το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα Κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ, δώστε μας την ε, διαβεβαίωση ότι θα μπορούν να σπουδάζουν οι φοιτητέ εκεί που θέλουν, στο εξωτερικό. Είναι απαράδεκτο να κινδυνεύει το πρόγραμμα Εράσμους. Ε, η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική είναι αυτοκτονική και παράλογη ε, καταστρέφει οτιδήποτε κρατικό και κινείται μόνο προς την ιδιωτικοποίηση. Ιδιαίτερως για τις ε, χώρες του Νότου είναι καταστροφικό. Όλος ο εκπαιδευτικός κόσμος στην Ισπανία είναι στο δρόμο για να προστατεύσει, να υπεραμεινθεί της ε, δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης ε, που απειλείται από την παρέμβαση της Τρόικας, από τις περικοπές. Το να κινδυνεύει το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα δυσχεράνει την κατάσταση και θα ε, ε, χειροτερεύσει τις ε, περικοπές, την αύξηση των διδάκτρων και θα οδηγήσει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους στην αύξηση των δανείων τους. Επίσης κινδυνεύει και η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Δημιουργούμε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, αυτό δεν είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε. Η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες παντού. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μάγερ. Η κυρία από το EFD. Πρόεδρε, το Έρασμος ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια και 3 εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Από το 2007 έως το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 3 δισεκατομμύρια ευρώ για το εράσμος. Όμως, η οικονομία συρρυκνώθηκε. Η ανεργία των νέων έφτασε στο 11,7%. Επίσης, ε, δίδονται μέσω του Εράσμου 300 ευρώ το μήνα που δεν καλύπτουν το βασικό κόστος ζωής. Αν προσθέσουμε και τα ταξιδιωτικά έξοδα, φαντάζομαι ότι θα πρέπει η οικογένεια να, να πληρώσει επιπλέον 5.000 ευρώ το χρόνο για να πέρα από αυτά που δίνει το Erasmus, ούτως ώστε να καλυφθεί το κόστος ζωής για το φοιτητή. Πόσες οικογένειες μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα στην περίοδο κρίσης. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας την την επίπτωση του έρασμου στην οικονομία την τελευταία δεκαετία και δεδομένου του ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν μόνο όσοι είναι πλούσιοι, θα πρέπει να το ξεχάσουμε, θα πρέπει να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Υπάρχουν άλλε προτεραιότητε που θα πρέπει να προωθήσουμε. Όσοι το θεωρούν απαραίτητο, θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη του τότε. Αντί να επιβάλλουν αυτό το βάρο στου ε, φορολογούμενου. Ευχαριστώ. Κύριε Αντρίεσεν, ο κύριο Σούσα Βάγνερ από του μη εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, το είδηση για το Εράσμους είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρή γιατί επηρεάζει την κατάρτιση ε, και τη διανόηση της στην Ευρώπη. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι πυλώνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό το λόγο το συντομότερο δυνατό ε, θα πρέπει να αναζητηθούν τα κατάλληλα κονδύλια από τα αντίστοιχε γραμμέ του προπολογισμού για να επιληθεί το πρόβλημα και να καθησυχαστεί η κοινή γνώμη κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, θα πρέπει οι αρμόδιοι ε, δημόσιοι λειτουργοί να προσέχουν πολύ όταν δημοσιοποιούν τέτοιου είδους ειδήσει. Ε, τα πρωτοσέλιδα ε, παραπέμουν σε μια ε, τρέλα, τρελή απόφαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Περνάμε στου ε, υπόλοιπου εγγεγραμμένου ομιλητέ. Ο κύριο Κουρία πρώτο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προηγούμενη συζήτηση αφορούσε τα 20 χρόνια της ενίας αγοράς την κάναμε γιατί η ενιαία αγορά είναι μία από τα βασικά ορόσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπήρχε η ενιαία αγορά, τότε δεν θα υπήρχε ενδεχομένως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έρασμος είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Για πολλού νέου, όχι μόνο, είναι η ίδια εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρί το έρασμο, για πολλού, δεν έχει κανένα νόημα η ενιαία Ευρώπη. Είναι πολύ ε, πιο σημαντικό για αυτού του νέου από την ενιαία αγορά. Γιατί η ενή αγορά ε, φυσικά έχει οικονομικά ωφέλη για τις περιφέρειές μας και για τις επιχειρήσεις μας. Αλλά το Εράσμος είναι κάτι άλλο. Είναι η θέληση των φοιτητών ε, να ανακαλύψουν την κουλτούρα άλλων χωρών, να βγουν έξω από τα σύνορά τους, να ακούσουν ανθρώπους που μιλάνε άλλη γλώσσα, που έχουν άλλη, άλλες συνήθειες και άλλες παραδόσεις, για να ανακαλύψουν, να βρουν, να ψάξουν και να ξανασυνθέσουν τη δική μας ταυτότητα. Έτσι γεννήθηκε η Ευρώπη όχι μέσα από τις συνθήκες, όχι μέσα από τη γραφειοκρατία, αλλά μέσα από την ε, πραγματική εμπειρία των πραγματικών ανθρώπων. Ε, χωρίς το έρασμους, ε, ίσως και η ενία αγορά θα είχε άλλο νόημα και άλλο πνεύμα. Επομένως, η αποδυνάμωση του Εράσμους θα σήμαινε αποδυνάμωση της ένωσής μας. Ο τίτλος αυτής της συζήτησης ε, είναι απόλυτα σωστός. Είναι σε κίνδυνο το Εράσμους. Υπάρχει κίνδυνο, ε, χωρίς το έρασμο, να περάσουμε σε μια άλλη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη δεσμευσή σα, και θα ήθελα και το Συμβούλιο να δεσμευτεί πραγματικά να βρεθούν τα λεφτά και να εγκριθούν. Γιατί αυτή η τρύπα που έχουμε εξαρτάται για την κάλυψή τη από, από τη θέληση των κρατών μελών. Η Ευρώπη βασίζεται ε, στις πλάτες αυτών που θέλουν να σπουδάσουν. Θα πρέπει λοιπόν να μην διαψεύσουμε τις προσδοκίες ε, τους. Καλή δουλειά στο Συμβούλιο και περιμένουμε μόνο καλά νέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις ε, τελευταίες εβδομάδες οι εφημερίδες αναφέρονται στο τέλος του Εράσμους. Είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε του ε, πολίτε ότι τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το Κοινοβούλιο Επικεφαλή ε, συνεργάζονται δραστηρία για το μελλοντικό προπολογισμό, ε, χωρί να θέτουμε σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα ενό προγράμματο όπω το Εράσμους. Το Εράσμους μας δείχνει τους κινδύνους των περικοπών και της λιτότητας πρέπει να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη ακόμα και σε περίοδο κρίσης είναι πρόθυμη να επενδύσει στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την οικονομική και την κοινωνική κρίση. Θα πρέπει να αποφύγουμε παρόμοια κατάσταση στο μέλλον γιατί παίζεται η αξιοπιστία των θεσμικών μας οργάνων. Πρέπει να βρούμε μια λύση για να δείξουμε το ενδιαφέρον μα για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρταση σε στιγμέ κρίση. Καλό το Συμβούλιο να συνεργαστεί λοιπόν με το Κοινοβούλιο και με την Κομισιόν προκειμένου να βρούμε μια λύση και να εξασφαλιστούν τα 90 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται. Σα ευχαριστώ και η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χάρη στο Εράσμους είναι μια θετική εικόνα. Αυτή τη στιγμή υποσκάπτουμε αυτή την εικόνα. Είναι μια στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολίτες, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ανησυχούν για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το πρόγραμμα αυτό όμως έχει συνεισφέρει στην θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των πολιτών της. Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, υπογραμμίσατε τα προβλήματα που υπάρχουν για το 2012 και για τη χρηματοδότηση του Ερασμού. Δεν μας δώσατε όμως απαντήσεις. Το ερώτημα που απευθύνουμε στα κράτη-μέλη όλοι μαζί είναι έχετε δει το θέμα της συνεισφοράς σας στη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει. Πέραν του Εράσμους, το θέμα της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των του Ταμείου Συνοχής ε, ε, είναι δραματικό. Ζητώ αυτόνομη χρηματοδότηση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα επιτρέψει να βγούμε, να γλιτώσουμε αυτές τις τρέλες αποφάσει των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Erasmus έχει τις, τα όρια του, αλλά είναι ένας από, ένα από τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χάρη σε αυτό οι νέοι εκτιμούν την Ευρώπη. Είναι ένα μηχανισμό που οικοδόμησε την Ευρώπη, την Ευρώπη τη συνεργασία και όχι του ανταγωνισμού εναντίον όλων. Εάν ε, τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχούσαν πραγματικά για το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, δεν θα συζητούσαμε εδώ του περιορισμού και τι δραστικέ περικοπέ των πόρων. Αλλά θα δρούσαμε συλλογικά για να δώσουμε περισσότερε υποτροφίε, ούτω ώστε το Erasmus να μην αφορά μόνο το 4% των φοιτητών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ήδη σημαντικές. Ε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες το χειρότερο θα ήταν να αντικαταστήσουμε το σημερινό σύστημα με ένα σύστημα δανείων. Το αποτέλεσμα θα ήταν να ξεκινούν οι φοιτητές ε, την επαγγελματική του ζωή με ένα επιπλέον φορτίο στους ώμους. Αν θέλουμε η Ευρώπη να βγει από την κρίση θα πρέπει να αυξήσουμε πολύ σημαντικά το επίπεδο κατάρτισης και έρευνας, να υπάρχει, να γίνει μια κολοσιαία προσπάθεια. Είναι δική μας ευθύνη. Όχι μόνο το πρόγραμμα έρασμος ε- να διασωθεί, αλλά να αναπτυχθεί και να ανταποκρίνεται στα δικηβεύματα της εποχής μας. Είναι επίσης να επεκτείνουμε αυτό το, αναγκαίο να επεκτείνουμε το πρόγραμμα στην ε, διαβίου ε, εκπαίδευση των εργαζομένων, ούτω ώστε να υπάρχει σε επίπεδο ένωσης ασφάλεια για τη δουλειά τους, για τη δουλειά των εργαζομένων. Το πρόγραμμα Εράσμους θα πρέπει να το υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια ε, για το μέλλον των νέων μας. Ε, ίσως μπορείτε να κόψετε ε, τους υπερμισθούς και τις υπερσυντάξεις, αυτές τις διογκωμένες συντάξεις των γραφειοκρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης θα μπορούσαμε να περικόψουμε τους μισθούς των ε, μεγάλων τραπεζιτών. Ε, το έρασμος αφορά τους νέους και προτάθηκε στον πρόεδρο Μπαρόζο, ε, προτάθηκαν κάποια πράγματα. Ε, προτάθηκαν τρόποι για να ε, εξασφαλιστεί αυτή η κινητικότητα των νέων χωρίς να είναι βάρος για τους γονείς τους. θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε με προγράμματα ε, όπου θα συμμετείχαν οι βιβλιοθήκες που θα δίνουν δανεικά βιβλία κτλ. Επίσης, μην ξεχνάμε και την αρχή της επικουρικότητας. Ας διευρύνουμε την ε, συμμετοχική βάση του Εράσμου. Ας δώσουμε ρόλο ε, και για προτάσεις και για παρεμβάσεις ε, στους νέους μας. Το Εράσμους είναι κάτι σημαντικό. Εμείς οι ευρωκριτικοί σκεπτικιστές υποστηρίζουμε το Εράσμους πολύ περισσότερο από τους υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θέλουμε να κρατήσουμε το Εράσμους γιατί είναι το μέλλον των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη το όρισε η Doris Πακ, έχουμε να εκφράσουμε μια ανησυχία για τις δραματικές ε, συνέπειες ε, τις οποίες θα, έχει, θα έχουν οι περικοπές σε λάθος τομέα, δηλαδή στην εκπαίδευση ενώ είναι σαφές πως εκεί πέρα έχουμε το ισχυρότερο όπλο κατά της κρίσης, της ανεργίας και οπωσδήποτε υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Ένα κομμάτι ευρωπαϊκής επιτυχημένης πολιτικής, όπως είπε ο κύριος Κουρία, που είναι εξίσου σημαντικά όσο η εσωτερική αγορά και το ευρώ και κινδυνεύει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί και ελπίζω να έχουμε καλό αποτέλεσμα και ελπίζω η Κομισιόν να μην επαναλάβει άλλες φορές δηλώσεις σαν αυτές της 15ης ε, Οκτωβρίου όπου είπε πως δεν μπορεί να εγγυηθεί τη χρηματοδότηση του Εράσμους γιατί δεν αναλαμβάνει το Συμβούλιο της Ευθύνης του. Απευθύνω έκκληση στο Συμβούλιο με όλους τους συναδέλφους εδώ πέρα πως η ευθύνη που έχουμε απέναντι στις με επόμενες γενναίες πρέπει να αναλυφθεί και με τρόπο επαγγελματικό. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Λεβαντόφσκι, εκπρόσωποι του Συμβουλίου, δύο μέρες πριν είχαμε μία συζήτηση για τον προϋπολισμό του 2013 και μεταξύ άλλων μιλήσαμε για τα προβλήματα που θα έχουμε του χρόνου με τις πληρωμές εάν το Συμβούλιο δεν δεχτεί την πρόταση της Κομισιόν και την ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για τον έρασμο θέλουμε να δούμε τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά. Ποιο είναι το μέλλον του έρασμου δηλαδή. Επειδή δεν έγινε αποδεκτή η θέση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου πέρσι. Γι' αυτό μία σειρά προγραμμάτων μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Ο κύριος Μαυρογιάννης μας είπε ότι αυτό δεν θα συμβεί, δεν θα υπάρχει πρόβλημα πληρωμών. Ε, αυτό μας ελέγχθηκε πέρσι, δεν το πιστεύουμε, λυπάμαι μας ελέγχθη ότι θα υπάρχουν αρκετά χρήματα και φέτος η Επιτροπή υπέβαλε διορθωτικό προϋπολογισμό 2 ε, δις ευρώ. Το θέμα θα πρέπει να επιληθεί. Θα πρέπει να δεχτούμε την πρόταση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Νίτρας για 1,5 λεπτό. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, szanowni Państwo, w okresie, kiedy Κυρίες και κύριοι, τη στιγμή που μιλάμε για θέματα απασχόλησης και απασχολησιμότητας, οι νέοι αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από τις άλλες ηλικιακέ ομάδες. Υπάρχει μεγάλη απειλή για το πρόγραμμα Έρασμος και η συμπεριφορά του Συμβουλίου δείχνει ότι φέρει μεγάλες ευθύνες. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουν οι νέοι τα προβλήματά τους. Εμείς λύνουμε τα δικά μας, αλλά δεν λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών της Ευρώπης. Αντιμετωπίζουμε μεγάλη κρίση και πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ότι μας χρειάζονται, χρειάζονται την Ευρώπη. Και αυτό το μήνυμα δείχνει επακριβώς ότι υπάρχει ε, μεγάλη αλληλεξάρτηση και θα ήθελα να πω στους Λαμασούρ και Λεβαντόφσκι ότι είμαι ευγνώμων γιατί περιμένουμε να εισακουστεί η φωνή τους. Διαφορετικά θα πεθάνει εν σιωπή το πρόγραμμα Ερασμός. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μικάλσκι, επέκρινε την Κομισιόν και τώρα η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να μιλήσουν με μία φωνή. Και χαίρομαι διότι υπάρχει συνεκτική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, ως προς τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την οδηγία 665 του 99 ορίσαμε τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει να εργάζονται οι μισθωτοί και εκεί υπάρχει και το θέμα της ελάχιστης θερμοκρασίας στον χώρο εργασίας. Δεν ξέρω, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει σωστή ε, θερμοκρασία ούτε σε αυτή την αίθουσα και μιλώ για τη φυσική θερμοκρασία, όχι την πολιτική. Κύριοι συνάδελφοι, θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Θέλω να σας ενημερώσω ότι περισσότεροι από 20 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και δεν είναι δυνατόν, ε, επειδή έχουμε ψηφοφορία στις 12, να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσει, οπότε θα ήθελα ε, να παρακαλέσω τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στην προηγούμενη ε, συζήτηση να δώσουν προτεραιότητα στους συναδέλφους τους. Παρακαλώ την Αντιπρόεδρο Ρομπέρτα Αντζελίλη πρώτα. Eh, Πρόεδρε, δεν μπορούν οι νέοι να καταβάλουν το τίμημα της οικονομικής ε, κρίσης. Υπάρχει μεγάλη οικονομική ε, κρίση και θα πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες και τις υπερβολικές δαπάνες. Αλλά δεν μπορούμε να αγγίξουμε τα ταμεία και τα προγράμματα που λειτουργούν. Δηλαδή, εν πρώτη στον ε, έρασμο, που δίνει δυνατότητες σε πολλούς νέους της Ευρώπης Πρόκειται για νέους που δεν έχουν ε, μεγάλες οικονομικές δυνατότητες ε, για κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε για να μπουν στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για έναν τόπο και χώρο εργασίας που είναι δύσκολος ε, και δύσβατος για τους νέους. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους νέους που προσμένουν κάτι από εμάς, που παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να τους πούμε ότι δεν θα αγγίξουμε το πρόγραμμα Έρασμος και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να τηρήσουμε αυτό το στόχο. Ε, ο συναδελφος Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το Εράσμους κατά κοινή παραδοχή όλων μας είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόγραμμα που είναι ταυτισμένο με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ως εκ τούτου, συζητώντας σήμερα για το αν αυτό το πρόγραμμα είναι σε κίνδυνο, για μια ακόμη φορά θέτουμε τους ίδιους μας σε αυτούς σε αφισβήτηση. Το ίδιο υπενθυμίζω κάναμε το προηγούμενο διάστημα και για το χώρο Σέγγεν, κάτι ανεπίτρεπτο. Θέλω λοιπόν, συνεχίζοντας τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, να ζητήσω από όλα τα νέα παιδιά όλους τους φοιτητές σε όλη την ευρώπη στις 33 χώρες που εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό να συνεχίσουν να κάνουν αιτήσει να είναι βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά θέλω επίση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στου διδάσκοντε και σε όλου εκείνου που εμπλέκονται στην εφαρμογή του προγράμματο οι οποίοι πολλέ φορέ και με προσωπικέ θυσίε φροντίζουν να πηγαίνουν όλα καλά γιατί υπόθηκε και προηγουμένω πολλέ φορέ οι πόροι από το εράσμου δεν επαρκούν. οι κυβερνήσει έχουν κάνει λάθη κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η ευρωπαϊκή επιτροπή για να δείξουμε ότι τα αυτονόητα δεν τα συζητάμε ξανά. αν στο μέλλον έχουμε μια τέτοια δυσάρεστη συζήτηση ξανά η συζήτηση δεν θα είναι για το αν το εράσμου έχει πρόβλημα θα είναι για το αν η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε Παπα-Νικολάου, η συνάδελφος Σίλβια Κώστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε και εκπρόσωπε του Συμβουλίου, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του προγράμματος Έρασμος οι 33 χώρες και τα 2,5 εκατομμύρια φοιτητών που είχαν τη δυνατότητα κινητικότητας προς αυτή την κατεύθυνση έχουν μεγάλες αμφιβολίες. Είναι αδιανόητο να τίθεται ένα αμφιβόλο η επιτυχία αυτού του προγράμματος τη στιγμή που είχαν, είχαν απορροφηθεί οι πόροι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συνολικό ε, πρόγραμμα Long Life ε, Learning αποτελεί το 0,7% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάμε για την επόμενη επταετία για μία αύξηση της τάξης του 65%. Μα είναι τερατώδες να αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει δέσμευση. Χαίρομαι διότι η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να λάβει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα πρέπει να μιλήσουμε με ενία φωνή για να μην γίνουν ευρωσκεπτικιστές και οι νέοι. Η κυρία Τσικάου. Το πρόγραμμα Έρασμος είναι ένα εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για κινητικότητα των νέων πέρα από τα αγαθά και τα κεφάλαια. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι στην περίοδο 14-20 θα πρέπει να υποβοηθήσουμε αυτό το πρόγραμμα με σημαντικές αυξήσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την υψηλή ανεργία σε επίπεδο νέων σε όλα τα κράτη-μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εκπαίδευσης ε, για τους νέους, μιλάμε για αύξηση του προγράμματος Έρασμος για τις ε, επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά να λάβουμε υπόψη και την συμπερίληψη των νέων μέχρι τα 35 χρόνια και να προωθήσουμε και την κινητικότητα στον τομέα των επιχειρήσεων, μιλώντας για τον έρασμο, πρόγραμμα έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς ε, και τη σημασία του προγράμματος και για τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στα παιδιά και στους νέους. Αυτοί οι οποίοι είναι αρνητικοί απέναντι στην ευρωπαϊκή συνεργασία λένε πως ε, δεν επαρκεί το πρόγραμμα Εράσμους για να γίνει επιτυχής η Ευρώπη. Μα τώρα εδώ πέρα έχουμε βήματα προς τα πίσω. Πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στην κινητικότητα. Γνωρίζουμε πως ε, η αγορά χρειάζεται ε, εκπαιδευμένους ε, εργαζόμενους και πραγματικά αυτό ήταν το όφελος του πολύ επιτυχούς αυτού προγράμματος. Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις στην εκπαίδευση ειδικά τώρα και είναι ανησυχητικό να κόβουμε αυτό το πράγμα. Θεωρώ πως ε, η Κύπρος δεν θα ήθελε να είναι η Προεδρία εκείνη η οποία θα στείλει ένα τέτοιο αρνητικό μήνυμα ειδικά εφόσον μπορεί να έχει και μια ιδιαίτερη ευθύνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με το πρόγραμμα Έρασμος ε, έχουμε ε, ένα πρόγραμμα υποτροφιών όπου μπορούν να προωθηθούν οι νέοι σε επίπεδο επιστημονικό αλλά και γλωσσικό. Εμείς οι νεότεροι βουλευτές, ευρωβουλευτές, χρησιμοποίησαμε αυτή την υποτροφία γιατί γνωρίσαμε πολλούς νέους που δεν θα είχαμε γνωρίσει εάν δεν μπορούσαμε να βγούμε στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι προνόμιο ε, για τα παιδιά των πλουσίων. Ρωτώ το Συμβούλιο και την Επιτροπή ποιος είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα πληγούν από αυτές τις περικοπές. Σε αυτή την περίοδο ανεργίας των νέων χρειάζεται ακόμα περισσότερο, χρειάζονται ακόμα περισσότερο αυτές οι υποτροφίες και ανταλλαγές, γιατί η Ευρώπη δεν θα αλληλοκατανοηθεί χωρίς το πρόγραμμα Έρασμους. Φερνάντες. Ε, χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανεργία των νέων είναι διπλή σε σχέση με τις άλλες ε, γενναίες. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα Έρασμος ε, βοηθά τους φοιτητέ σε ακαδημαϊκό και επιστημονικό επίπεδο και ενισχύει και τις δυνατότητες εξέβρεσης εργασίας. Γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο έχει αναλάβει δεσμεύσεις. Θα ήταν απαράδεκτο λοιπόν ε, να έχει ως σύνθημα το Συμβούλιο «Δεν πληρώνουμε». Θα πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του. Θα πρέπει να γνωρίζει ότι πρόκειται για θέμα εμπιστοσύνης. Είναι ένα κατά προτεραιότητα πρόγραμμα, έτσι ώστε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα να συνεχιστεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες για τις σχετικές ε, πληρωμές. Παλιαδέλη. Κυρία Πρόεδρε, ε, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα ότι μετέχω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση ε, ακριβώς γιατί στα 25 χρόνια του πετυχημένου αυτού προγράμματος συζητούμε, αναρωτιόμαστε αν πρέπει να το συνεχίσουμε ή όχι. Θεωρώ ότι τα πιο πετυχημένα προγράμματα της Ευρώπης εξαντλούν τα αποθέματά τους ακριβώς γιατί είναι πετυχημένα. Είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών να στηρίξουν τα πετυχημένα προγράμματα γιατί στηρίζουν έτσι το μέλλον της Ευρώπης. Χαίρομαι ιδιαίτερα ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου υποστηρίζει ένθερμα όχι μόνο τη συνέχιση του προγράμματος, κυρίως όμως το μέλλον του και επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ίδιο αυτό πρόγραμμα και στον επόμενο προϋπολογισμό. Ευχαριστώ ευχαριστώ και εγώ πολύ ο συνάδελφος Ράνστορφ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ένα ε, απλό ερώτημα που σχετίζεται με μια διατριβή που είχα διαβάσει τη δεκαετία του 80 όταν δούλευα στην Ακαδημία Επιστημών. Τότε ένα 35% του ΑΕΠ και της αύξησής του προέρχονταν από την εφαρμογή της έρευνας και της ανάπτυξης. Έκτοτε το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κιόλας. Και τι κόβει εδώ πέρα η Κομισιόν την έρευνα και την ανάπτυξη. Δηλαδή το πιο χρήσιμο εργαλείο για να ξεπεραστεί η κρίση. Και πρέπει να ακούσουμε από την Κομισιόν γιατί ακριβώς υπονομεύουμε αυτό το δυναμικό ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Το πρόγραμμα Έρασμος ε, αντικατοπτρίζει την κατάσταση του προϋπολογισμού. Μεγάλη ανευθενότητα των ε, δεσμεύσεων που, στις οποίες δεν ανταποκριθήκαμε και δηλώσεις πολύ θεματικές σε κάθε συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά καμία ανταπόκριση ως προς, προς τις ε, πληρωμές. Ο κύριος Λεβαντόφσκι επεξήγησε την κατάσταση στην ουσία σέρνουμε έναν προϋπολογισμό και μιλάμε για ένα έλλειμμα που είναι της τάξης των 130 δις. Δεν ήμασταν σε θέση να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας. Γι' αυτό η Επιτροπή Προϋπολογισμών και ιδιαίτερα ο κύριος Λαμασούρο Πρόεδρος έκανε μία δήλωση στον τύπο μιλώντας ε, για την κατάσταση του προγράμματος ε, Έρασμος, θεωρώντας ότι δεν θα πρέπει να επαπειληθεί αυτό το ε, πρόγραμμα. Μπόρις. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σύντομα, μιλάμε για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ε, γύρω στα 2,5 εκατομμύρια φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εράσμους και μας κοιτάνε αυτή τη στιγμή, αναμένουν το εάν θα είμαστε αρκετά αποφασισμένοι να τους δώσουμε άλλη μια ευκαιρία για περισσότερη ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το Εράσμους εάν, θέλουμε, εάν θέλει κανείς να βελτιώσει τα προσόντα του. Και αυτές είναι εμπειρίες που συνοδεύουν τους νέους σε ολόκληρη τη ζωή τους. Και ελπίζω λοιπόν η δραστηριότητά σας να έχει αποτελέσματα σε αυτή και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Γνωρίζω επίσης πως σας αρέσει ο αθλητισμός, γι' αυτό έχω να σας δώσω και ένα συμβολικό μπλουζάκι με το όνομά σας και μετά το χθεσινό αγώνα θα ήθελα να είστε κι εσείς ε, τόσο αποτελεσματικό όσο και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στον αγώνα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι το μόνο που λειτουργούσε θετικά στην Ευρώπη ήταν το ε, πρόγραμμα Έρασμος. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι και στην ε, περιοχή ε, των Αστουριών είχαμε υποδεχτεί την ε, Επίτροπο Ρέντινγκ και θεωρήσαμε ότι το πρόγραμμα Erasmus είναι ένα από τα λίγα προγράμματα τα οποία είναι επιτυχημένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν τόσο σύντομος. Ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους που δεν πήραν το λόγο ότι μπορούν να καταθέσουν γραπτή δήλωση που δεν θα υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία προσαρτάται στα πρακτικά της ε, συζήτησης. Και θα ήθελα τώρα ε, να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Λεβαντόφσκι. Madam President, colleagues, thank you for your real Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για αυτή την αφοσίωση, την πολύ επίκαιρη ε, αφοσίωση στην προσπάθεια να σωθεί το έρασμος. Είναι η στιγμή να χτυπήσει το καμπανάκι. Ευχαριστώ επίσης που μου θυμήσατε με το δώρο σας ότι ο Λεβαντόφσκι κατάφερε να βάλει γκολ για τη Ρεάλ Μαντρίτ. Όμως αυτό είναι μια ευκαιρία να δούμε τι κρύβεται πίσω από τα νούμερα. Καμιά φορά είναι απαραίτητο να βλέπουμε τι, είναι, βρίσκεται πίσω από τα νούμερα του προϋπολογισμού. Είναι πολύ εύκολο να μειώσει κανείς τα ποσά πάνω στα χαρτί, αλλά όταν βλέπει τους φοιτητέ του Εράσμους είναι πιο δύσκολο ή όταν βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πίσω από τα νούμερα, επιχειρήσεις που είναι σε απελπιστική θέση σε μια περίοδο περιορισμού των πιστώσεων, δεν είναι πολύ εύκολο μειώσουμε τα νούμερα. Αυτό και συνέβη με το Εράσμους. Ξεκίνησε με νομίζω ένα μικρό ποσό το 1988, 18 αν δεν κάνω λάθος εκατομμύρια ευρώ και πάνω από 4.000 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 33, σε 33 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνυπογράψει το χάρτη του Εράσμους και αυτό δεν είναι απλώς ε, ένας τρόπος να φανεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το χρειαζόμαστε τώρα, τη χρησιμότητα των θεσμικών μας οργανών. Όπως σας εξήγησα η κατάσταση έχει ως εξή. Ε, έχετε την ε, διαβεβαίωσή μου, θέλω να σας διαβεβαιώνω και νομίζω ότι το στηρίζει αυτό και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Μαυρογιάννης, ότι οι φοιτητές που φέτος χρηματοδοτούνται από το Εράσμους και στις αρχές του 2013 επίσης δεν θα διακινδυνεύσουν. Όλα θα πραγματοποιηθούν επειδή έχουμε στείλει χρήματα στους εθνικούς οργανισμούς 33 χωρών. Αυτό που διακυβεύεται, ε, ε, ιδίω αν επωφεληθούμε ε, από τα ποσά του 2014 για να καλυφθούν οι ανάγκες του 2012 και τα επιπλέον αιτήματα είναι η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα επηρεάζει κυρίως τους φοιτητές που προέρχονται από, μειονεκτικά, ε, από μειονεκτικές ε, οικογένειες, τους φτωχότερους φοιτητές. Χρειαζόμαστε λοιπόν την δέσμευσή σας, την αφοσίωσή σας. Μην ξεχνάμε ότι το εράσμος είναι ένα κομμάτι μόνο της όλου προγράμματος για τη διαβίου μάθηση. Υπάρχει και το πρόγραμμα Marie Curie για νέους ερευνητές που επίσης κινδυνεύει αν δεν έχουμε επιπλέον 100 εκατομμύρια φέτος. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Σε μια στιγμή που ξεκινάμε μια μάχη για το μέλλον μέχρι το 2020. Δεν ισχύει ότι αυτά τα πρόγραμμα θα επηρεαστούν. Αυτό είναι το, το πιο αυξανόμενο κομμάτι του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από 15 σε 18. Ε, αλλά αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να διαβεβαιώσουμε τους θητητές ότι το 2013 δεν θα επηρεαστούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεβαντόφσκι και σας ευχαριστώ και για την δουλειά που έχετε κάνει τώρα. Ο κύριος Μαυρογιάννης, ο Υπουργός ε, εξ της Κυπριακής Προεδρίας. Παρακαλώ καθίστε ε, λίγο ήσυχα. Honourable members, thank you very much for this debate. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ, πολύ. για αυτή τη συζήτηση. Θα ακολουθήσουμε τις προτάσεις του κυρίου Σβόμποντα, όπως επίσης και όλες τις ανησυχίες και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν. Τα έχω σημειώσει, θα μεταφέρω και στα κράτη-μέλη και στο Συμβούλιο. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι συμμεριζόμαστε την ε, άποψη ότι η κινητικότητα των φοιτητών και το Εράσμους είναι βασικό, βασικά ε, μέσα για τη νέα γενιά. Μπορείτε να κάνετε λίγο περισσότερη ησυχία δείχνοντας σεβασμό στον ομιλητή και στους συναδέλφους. Uh, Έλεγα ότι συμφωνούμε κι εμείς ότι η κινητικότητα των φοιτητών ότι και το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους είναι κομμάτι του οραματός μας για το μέλλον και θεωρούμε ότι δίνει νόημα στην Ευρώπη. Όσον αφορά τα κονδύλια του 2012 το Συμβούλιο, όπως έλεγα και προηγουμένως, θα συνεχίσει γρήγορα την εξέταση του σχεδίου προπολογισμού 6 που προτείνει η Κομισιόν και θα αναλύσουμε τυχόν ελλείψεις κονδυλίων που έχει εντοπίσει η Επιτροπή στον τρέχοντα προπολογισμό για όλα τα προγράμματα συμπεριλαμβανομένης και της διαβίου μάθησης συμπεριλαμβανομένων και των βασικών στοιχείων Εράσμους και Μαρή Κιουρί. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευθεί αποφευχθεί η κατάσταση που όλοι φοβάστε. Δηλαδή να μην μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να εξασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος Εράσμους. Όσον αφορά το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μόλις ξεκίνησαν μια διαδικασία στην διαλλαγή με σκοπό να ευρεθεί μια συμφωνία στο επίπεδο κονδυλίων και πιστώσεων στο επόμενο προπολογισμό και βεβαίω εδώ συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα διαβίου όπως σας έλεγα προηγουμένως συμπεριλαμβανομένου και του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου 2013-2020 γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων όμως η εντύπωσή μου είναι ότι το Εράσμου δεν κινδυνεύει. Δεν πρόκειται να, επιτρέψει, να, το αφήσουν να συμβεί αυτό. Υπάρχει μεγάλη ε, αφοσίωση στο Εράσμου. Σε ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Στις 12 ακριβώς θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή λοιπόν.